που πήγαν να διαμαρτυρηθούν κατά των πολιτικών παιχνιδιών των ρουμανικών κομμάτων και ζήτησαν να, γίνουν σεβαστές οι ουγγρικές κοινότητες. Ο κ. Πόζας έχει το λόγο για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε.